η συζήτηση. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο στις 12 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 9. Ε, τα, η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί, ε, διατίθεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και λύεται η συνεδρία.